Uh, dear colleagues, uh, Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Έχουμε ακόμα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος εισηγητής έχει το λόγο. Συνάδελφοι, έχουμε ακόμα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Τα αποτελέσματα λοιπόν τη ε, ψηφοφορίας. Ο κ. Λάζαρος Λαζάρο λοιπόν υπέρ 19 ψήφοι, κατά μία ψήφος, αποχέ μία. Λέω μπριγκάτ υπέρ 11 ψήφοι, κατά 9, Αποχέ μία. Ζωάβ Φιγκρέρο 19 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και δύο αποχές. Σας ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή στην ακρόαση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σαρβάμα, τον εισηγητή μας, ο οποίος και θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης για τις πιθανές εξελίξεις και προσαρμογές στο εφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην ε, εξέταση του προπολογισμού ε, θα υπόκειται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του προπολογισμού. Να καλωσορίσω λοιπόν την Γενική Γραμματεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπό τη και θα δώσω πάρα αυτά το λόγο στον κύριο Σαρβάμα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ναι, όντω, μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εισηγητή τη γνωμοδότηση αυτή εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Το θέμα λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια πολύ σημαντική είναι η έκθεση του κ. Φερχόφστα της Αρμόδιας Επιτροπής και ελπίζω ότι η γραμματότησή μας θα μετρήσει στη τελική ανάλυση. Θα σας παρουσιάσω εν συντομία τις βασικές τρεις ιδέες που περιλαμβάνονται στην γνωματοδοτησή μου. Καταρχάς, ελπίζω ότι εξετάζοντας τις τρέχουσες εξελίξεις και προσαρμογές στο βαθμό που είναι δυνατές φυσικά στο τρέχον θεσμικό πλαίσιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα, μα όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην διαδικασία του προπολογισμού θα υπόκεινται. Και αυτό φυσικά δεν είναι μόνο θέμα κοινή λογική, αλλά αποτελεί και την ουσία, αν θέλετε, της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό αποτελεί αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να υπόκεινται στο δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει ότι και η Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο θα πρέπει να υπόκειται στον έλεγχό μας. Τέλος. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και την αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού κανονισμού προκειμένου να διευκρινιστούν οι στόχοι της διαδικασίας ε, απαλλαγές. Και θα πρέπει πιο σημαντικό να ορίζονται και οι κυρώσεις οι οποίες θα επιβάλλονταν σε περίπτωση που δεν ήταν σεβαστός, σεβαστή διαδικασία χωρίς της απαλλαγής. Και τρίτος, τρίτον, προτείνεται και αυτό είναι κάτι που μας απασχόλησε και σήμερα το απόγευμα και μάλιστα μας έχει απασχολήσει και σε άλλες περιπτώσεις με πιο οδυνηρό τρόπο, βρισκόμαστε σε μια θέση στην οποία δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά το διορισμό μελών του Ελληνικού συνεδρίου. Όσο έχει σήμερα η συνθήκη, είναι υπερβολικά σαφής φυσικά θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι η ερμηνεία του Συμβουλίου είναι πλέον ορθή. Για το λόγο όμως αυτόν ακριβώς θα πρέπει να διευκρινιστεί το πώς έχουν τα πράγματα. Και έτσι, όπως είπα και στην αρχή, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Ένωσης μας παίρνουν στα σοβαρά όταν λένε ότι εξετάζουμε και ελέγχουμε τις δαπανές του Ευρωπαϊκού Πολεπολογισμού. Και στο πλαίσιο αυτό είναι βασικό, βασικός φορέας του Ελεκτικό Συνέδριο. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρούμαστε εισαξί και σε ό,τι αφορά την, ε, το διορισμό των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου. Και άρα, συνοψίζοντας, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να λάβει υπόψη δεόντως τις αποφάσεις που λαμβάνει το κοινοβούλιο μας. Και ασφαλώς είναι καθήκον της Επιτροπής μας να εξετάζει τους υποψηφίους όπως και πράξαμε σήμερα με τους τρεις υποψήφιους αυτούς. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση, στο σχέδιο γνωμοδότησης και με χαρά να ακούσω ενδεχομένω τι ερωτήσει σα σε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόγγεν έχει ζητήσει το λόγο. Χαιρετίζω, λέει ο κύριος Βόγγεν, <clears throat> την χρονοδότηση αυτή, όπως πάντα βέβαια είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη Έχω κάποια σχόλια και κάποια ερωτήματα για αυτήν την γνωμοδότηση. Ε, Φυσικά η σοσιαλιστική ομάδα, όπως και οι άλλες πολιτικές ομάδες, θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να υπάρξει διαφάνεια, λογοδοσία και σωστός ε, έλεγχος για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναρωτιέμαι απλώς για τις παραγράφους 2 και 3 τι ακριβώς εννοείται εκεί. Λέτε, ορθά, ότι υπάρχουν κάποια θεσμικά όργανα που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται από την διαδικασία ελέγχου και λέτε ότι λόγω αυτού θα πρέπει να υπάρξει μια προσαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο συνθήκης. Πρέπει να αλλάξουμε τη συνθήκη, είναι τεχνικές αλλαγές ή πρέπει να υπάρξει πραγματικά αναθεώρηση των συνθήκων. Θέτω αυτό το ερώτημα γιατί αυτό είναι μια γνωμοδότηση προς την Συνταγματική Επιτροπή και ο λόγος που κάνω αυτή την έκθεση είναι για να δουν αν στο μέλλον <clears throat> θα χρειαστεί να υπάρξει μεταρρύθμιση των συνθήκων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μας να διευκρινίσουμε αν απαιτείται κάποια τροποποίηση των συνθήκων ή όχι. Η άλλη παρατήρησή μου αφορά την παράγραφο 9, ιδίω εκεί που αναφέρονται οι κυρώσεις. Και ξέρω ότι η Επιτροπή μας θέλει να εξασφαλίσει ότι γίνεται σωστός έλεγχος, ότι όλα τα θεσμικά όργανα υπόκεινται σε αυτόν τον έλεγχο και αν δεν ε, συνεργάζονται κάποια θεσμικά όργανα, όπως το παρελθόν, θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να τα ενθαρρύνουμε για να συνεργαστούν. Δεν ξέρω βέβαια αν εδώ η κυρώση είναι το πιο ε, πρόσφορο μέσο για να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ίσως μπορούμε να μιλήσουμε για ένα πακέτο μέτρων, μια σειρά κινήτρων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θεσμικών οργάνων που πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο. Και τέλος θέλω να πω κάτι για την παράγραφο 6 όπου αναφέρεται το, τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και ο ρόλος του σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το τι θέλει να κάνει η Συνταγματική Επιτροπή αν θέλει να εξετάσει χωριστά τις, ε, τους αποκεντρωμένους φορείς ή αν θέλει να τους αντιμετωπίζει από κοινού. Γιατί αν τις αντιμετωπίζει από κοινού αυτό σημαίνει ότι μειώνεται η δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει τα θέματα αυτά και γι' αυτό θα ήθελα διευκρίνηση για την παράγραφο Στη Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Πέτρη τον εισηγητή για το σχέδιο γραμματοδότησης. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, αυτά είναι ούτως ή άλλως τα αιτήματά μας που χρονολογούνται από μακροχρόνου. χρόνου ούτως ή άλλως. Σύμφωνα λοιπόν με τη γενική προσέγγιση. Ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζω και ένα δίλημα όσον αφορά την έκθεση Φερχόφστατ. Ε, διάβασε το κείμενο προσεκτικά. Αν δείτε τι προτείνει, προτείνει μια άλλη, μια διαφορετική Ευρωπαϊκή Ένωση με Υπουργό Οικονομικών, με σημαντικέ αλλαγέ όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, άλλη αντιμετώπιση των χωρών της Ευρωμάδας, έμφαση στον κοινωτικό προπολογισμό, στον ενωσιακό προπολογισμό, ε, στους ίδιους πόρους, τη φορολογία, επενδύσεις, αυξημένος ρόλος της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζής Επενδύσεων, της ΕΚΤ και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος. Το πώς θα λειτουργεί η Ένωση όσον αφορά τον προπολισμό και τον ελεγχό του. Το δίλημα <laughs> λοιπόν είναι το εξή. Δεν συμφωνούμε καμία με αυτέ τι προτάσει. Ε, και είναι εκ των πραγμάτων δύσκολο να σχολιάσει κάτι κανεί με γνωμοδότηση τη στιγμή που δεν συμφωνεί, αλλά ήθελα να περιπτώσει να τονίσω αυτή την κατάσταση. Αν βρούμε τρόπο, καλύτερο τρόπο να εξασφαλίζουμε πόρους και να τους δεπανούμε με πιο αποδοτικό τρόπο, τότε πρέπει και ο έλεγχος του προπολισμού αλλάξει και αυτός και ίσως ο ρόλος μας να γίνει πολύ πιο σημαντικός στο μέλλον. Όχι μόνο για το καλό του προπολισμού, αλλά και για τη λογοδοσία των θεσμικών οργάνων. Και αυτό ακριβώ πρέπει να συζητήσουμε με τα άλλα θεσμικά όργανα. Το αν δηλαδή μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτούμε θα 100% πριν πόρου. πόρους. Μετά να δούμε το θέμα της λογοδοσίας. Όπως είπα, είναι θέματα τα οποία διαφεύγουν, εκφεύγουν το πεδίο του προπολισμού. Οπότε δεν ξέρω αν με τη γνωμοδότησή μας θα μπούμε στη γενική συζήτηση ή θα αναφερθούμε μόνο στα πολύ συγκεκριμένα και τα επιμέρους. Αν θα αφήσουμε δηλαδή τα, ε, την Επιτροπή συστηματικών Υποθέσεων να συζητήσετε ουσιαστικά και τα μεγάλα. Πρόεδρο, θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Όχι. Κύριε Σερβαμά, ο εισηγητή. Παρακαλώ. Ναι, να σου πω. Πρώτον, ε, ευχαριστώ για τα σχόλια. παρέλειψα να αναφέρω στην εισαγωγή μου ότι βέβαια είναι αυτονόητο ότι αν μπορούμε να βελτιώσουμε το κείμενο είμαι ανοιχτό σε προτάσεις. Οπότε είμαι όλο αυτιά. Αν υπάρχουν προτάσεις, τροπολογίες. Όσον αφορά τον Ντένις, τον κύριο Ντεγιόγκς. Ναι, αναφέρθηκε σε γενικότερα ίσως και φιλοσοφικά ζητήματα. Όντως αυτή τη στιγμή έχει θερμολογηθεί η σύνολο εξελίξεων που δεν ξέρουμε πού θα βγει, όπως λέμε. Αλλά ό,τι είναι να γίνει, μπορεί να γίνει και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ξέρω, μετά από ένα ή δύο χρόνια η κατάσταση μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων στον προπολισμό ε, μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι θα ήταν μάλλον δύσκολο να αναφερθούμε τώρα στις λεπτομέρειες για να απαντήσω στο ερώτημά σας. είναι πραγματικά, το, το ξανασκέφτομαι τώρα, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ασχοληθεί κανεί με την τελευταία λεπτομέρεια και αυτό όλο μαζί αποτελεί μια πρόκληση. Άλλωστε, πώ να προβλέψει κανεί και το μέλλον. Γι' αυτό εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν θέλω να επισέλθω στι λεπτομέρειε, το ξαναλέω. Ούτε θα ήθελα να γίνει αυτό με τι τροπολογίε ε, έω την επόμενη Τρίτη. Το σκέφτηκα πάντως. Ε, και η θέση μου είναι αυτή πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, αν θέλετε κάτι άλλο, τι να σας πω. Ευχαρίστως. να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε το κείμενο της γνωμοδότησης να γίνει πιο συνεκτικό, πιο λογικό. Πάντως, στη φάση αυτή είναι δύσκολο να πει κανείς κάτι περισσότερο. Σοβαρά τον Τέρικ. και τα μάλλον επικριτικά του σχολείου. Στην παράγραφο 9. Εγώ να σα πω τι, τι είχα στο μυαλό μου. Έχουμε, ξέρετε, απογοητευτεί ξανά και ξανά. Τόσες φορές. Ε, είναι πολύ απλό έτσι. Το λέω, το λέω έξω από τα δόντια. Έχουμε απογοητευτεί τόσο πολλές φορές που ήθελα πραγματικά να, να, να ξυπνήσω τον αναγνώστη. Πιστεύω προσωπικά ότι καλό θα είναι να βγούμε έξω με ένα χειρό μήνυμα, με μια αυστηρή γνωμοδότηση, αλλά βεβαίως ταυτόχρονα να είμαστε και προσεκτικοί. Ε, αν είναι, δηλαδή, να προτείνουμε κάτι, δεν μπορούμε να προτείνουμε κάτι το οποίο δεν στέκει, τότε αυτό ακυρωνόμεθα. Όμως, ε, χρειαζόμαστε σίγουρα κάποιου ορισμού κάποιες συγκεκριμένε θέσει. Πρέπει κάτι να πούμε. Πρέπει να πούμε ότι αν αυτό είναι ο ρόλο μα, αν αυτό μα ζητάτε να κάνουμε, να του λέμε ότι θα το κάνουμε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Το σε τι βάθος θα πάμε, σε πόσες λεπτομέρειες θα επισέλθουν, αυτό δύσκολα απαντάτε. Αλλά στο μυαλό μου είχα κάτι γενικό, αυτό θέλω να πω. Ας πούμε, εδώ λέει θέσπιση συγκεκριμένων ε, κυρώσεων στην περίπτωση μη συμμόρφωση κλπ. Πρέπει να προσδιοριστεί αυτό. Τώρα στις παραγράφους 1, μάλλον 2 και 3, 2 και 3, Το κλειδί βρίσκεται μάλλον στην παράγραφο 3. Λέμε ότι το γράμμα της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήστε του πνεύματος κλπ. τι άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και εδώ ο καθένας θα μπορούσε να δώσει το δικό του ορισμό, να ερμηνεύσει κατά δοκούν ποιο είναι το πνεύμα και ποιο είναι το γράμμα. Και όμως σκοπός μου ήταν να καταδείξω την απόκληση, τη διάσταση μεταξύ των δύο. Γιατί, ωραία, δεν συμβαίνει πάντοτε, δεν συμβαίνει κάθε φορά, αλλά συμβαίνει συχνά. Οπότε, κάτι πρέπει να γίνει. Το εύλογο ερώτημα και πάλι είναι να, να προτείνουμε τι, τι, να ξαναγράψουμε τις συνθήκες ε, δεν, νομίζω. <laughs> Δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν ρεαλιστικό. Όμως, ας σπρώξουμε όσο μπορούμε. Αυτή είναι και η τελική μου θέση. Και ας το κάνουμε αυτό σε κάθε παράγραφο. Όπου έχουμε κάτι να πούμε. Αν, όπου, αν και εφόσον δηλαδή έχουμε κάτι συγκεκριμένο να προτείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα υπενθυμίζω την προθεσμία των τροπολογιών στις 13 Σεπτεμβρίου και η έγκριση θα είναι στην 12 Οκτωβρίου. Ε, και μετά θα ακολουθήσει η έγκριση στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ. Πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η, αποστολή της Επιτροπής μας στην Ιορδανία και το Λίβανο. Decided to organize a mission to Jordan and Lebanon, which are the countries hosting the highest number of Palestinian refugees over 2 million in Jordan and half a in uh, Lebanon. The mission will take place uh, uh, from 20 until 23 Σεπτεμβρίου σε δύο εβδομάδες και θα περιλαμβάνει οκτώ μέλη μας μαζί με την ε, πρόεδρό μας, την ερήτημο πρόεδρό μας και έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα προετοιμασίας του προγράμματος της αποστολής μας. Έχουμε και εκπροσώπους της Διτζινία. Ε, ε, καλώς ήλθατε. Κύριε Άντερσον, χαίρομαι λοιπόν για την παρουσία σας. Και ίσως θα ήταν τόσο πιο σωστό να σας δώσω αμέσω το λόγο. Γιατί μπορούμε να έχουμε αυτή την ε, συζήτηση και θα περάσουμε σε κάποια σε κάποια ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συμμετάσχουμε σε αυτή την ε, αποστολή και <clears throat> θα έχουμε περαιτέρω συναντήσεις με την κυρία Γκρέσλε για τα θέματα αυτά. Η τελευταία μας συνάντηση ήταν στις 31 Αυγούστου. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον φορέα μας και μετά θα δώσω την κυρία Φάμπιαν το λόγο για να σας πει περισσότερα για την Ιορδανία και τον Λίβανο. Έχουμε και ένα συνάδελφο, μία συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού, αν θέλετε περισσότερα στοιχεία. Όπως ξέρετε, εμείς λειτουργούμε στις πέντε χώρες της περιοχής, Ιορδανία, Συρία, Λίβανο, την Δυτική Όχθη και την Λόριδα της Γάζας. Περίπου ένα δισεκατομμύριο ε, δολάρια το χρόνο είναι ο προϋπολογισμός και δίνουν τις βασικές υπηρεσίες για τα, το μεγαλύτερο μέρος των 5 ε, εκατομμυρίων προσφύγων στην περιοχή. Η ΟΥΡΑ εξασφαλίζει τη βασική παιδεία σε περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά. Έχει περίπου 150 κλινικές που λειτουργούν. Πρόκειται για ένα μεγάλο σύστημα το οποίο δίνει βασικές υπηρεσίες σε περίπου 5 εκατομμύρια άτομα στην περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολή μέσα στο πλαίσιο αυτό των προσφύγων. Όπως είδατε στον πόλεμο της Λωρίδας της Γάζας, ήταν από τους λίγους φορείς που ήταν ήδη επιτόπου και έδωσε άμεση βοήθεια <clears throat> και αρρωγή στα άτομα που είχαν ανάγκη στην ε, Λωρίδα της Γάζας. Ως ε, εκπρόσωποι λοιπόν της Κομισιόν μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας και θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ρόλο αυτού του φορέα στις πέντε αυτές περιοχές και όπως ξέρετε είναι ο μόνος φορέας του ΟΗΕ που δίδει ανεξάρτητα, προσφέρει ανεξάρτητα τις υπηρεσίες του. 90% του προσωπικού του, του φορέα αυτού είναι λειτουργικό προσωπικό, είναι δάσκαλοι, είναι γιατροί, είναι νοσοκόμοι, νοσοκόμες που εργάζονται σε αυτές τις περιοχές και στα κέντρα εκπαίδευσης και τα υγειονομικά κέντρα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει ο προϋπολογισμός. Έχουμε έχουν πάρα πολύ μεγάλες ε, δυσκολίες να αλλάξουν τον προϋπολογισμό αυτών των ε, ενεργειών, γιατί το 80% του προϋπολογισμού είναι για μισθοδοσία του λειτουργικού προσωπικού. Ε, χρηματοδοτούμε αυτό το, τους φορείς του Ηνωμένου, των με τρεις τρόπους. Καταρχήν με ένα βασικό ταμείο που παρέχει παιδεία και κοινωνικές υπηρεσίε από το προπολογισμό προγράμματος αυτού του φορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε αυτήν την συγχρηματοδότηση από το φορέα αυτό, αλλά επίσης δίνουμε χρηματοδότηση από δύο άλλους διάβλους που είναι το Ταμείο Έκτακτης Βοήθειας και συγκεκριμένα σχέδια τα οποία ζητούν οι επιτόπου φορείς. Αν συνενώσετε όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει περίπου 120 ε, εκατομμύρια το χρόνο σε αυτόν τον φορέα και μαζί με τα κράτη-μέλη όλα αυτά είναι περίπου 40% του συνολικού του προϋπολογισμού του φορέα αυτού. Του του έχουμε προβλήματα γιατί ο προϋπολογισμός ο συνολικός είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο για την συνδυματοδότηση των βασικών τους υπηρεσιών. 660 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τις βασικές υπηρεσίες και κάθε χρόνο έχει ένα έλλειμμα περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός ο φορέας είναι πολύ δύσκολο να καλύπτεται <clears throat> αυτό το χρηματοδοτικό χάσμα κάθε χρόνο και επανερχόνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν ξέρουν πώς να καλύψουν τη μισθοδοσία των τελευταίων μηνών του χρόνου, πώς να καθίσουν τα σχολεία ανοιχτά στη Γάζα ή στην Ιορδανία δεν υπάρχει λοιπόν επάρκεια προπολογισμού για να καλυφθεί αυτό το κενό. Κάθε, έτος του χρόνου, κάθε τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητείται να βοηθήσει περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη πίεση στον φορέα αυτό γιατί έχει αυξηθεί ο πληθυσμό των προσφύγων και έχει μειωθεί η βάση των χορηγών. Κάποιοι χορηγοί δίνουν όλο και λιγότερο στο φορέα αυτό. Κάποιες χώρες του κόλπου έχουν σταματήσει την υποστήριξή του στο φορέα αυτό και τώρα είμαστε στις 5 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά τελειώνουν τα λεφτά ήδη για το 2016. Μας είπαν ήδη χθε λοιπόν ότι αν δεν δώσουμε πρόσθετα α, κονδύλια για τη χρηματοδότηση των κύριων ενεργειών της ΣΟΥΡΑ, από τον Οκτώβριο δεν θα μπορούν να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο επανέρχεται σχεδόν κάθε χρόνο. Έχουμε τρία κέρια μηνύματα λοιπόν να σας δώσουμε και θα χαιρόμαστε αν μπορούσε αυτή η, η, η αποστολή σας να μας βοηθήσει να τα κάνουμε γνωστά σε όλους. Φυσικά εμείς υποστηρίζουμε την Ούνρα για το πολύ καλό της έργο, αλλά ζητούμε να συνεχιστεί και η εσωτερική διαδικασία μεταρρύθμισης, να γίνει πιο διαφανής ο προϋπολογισμός τους, να εστιάζουν περισσότερο στις βασικές υπηρεσίες που παρέχουν και όχι να διευρύνουν την δραστηριότητά τους σε άλλους τομείς ενέργειας. Επίσης να διευρύνουν τη βάση χορηγών τους. Δεν είναι φυσιολογικό να είναι ο χορηγός τελευταίας καταφυγής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες του Περσικού κόλπου θα έπρεπε να ζητηθεί να δώσουν περισσότερα χρήματα. Ε, χώρες όπως ο Καναδάς δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ, ούτε η Νορβηγία. Αντί λοιπόν να ζητείτε πάντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ζητηθεί να, καλύψει το, να καλύψουν το κενό αυτό και άλλες χώρες. Το τελευταίο και κέριο μήνυμα είναι, είναι ότι θέλουμε να ζητήσουμε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ψηφίσει για την ε, ε, καταβολή περισσότερων ποσών στον φορέα της ούρα. Όπως ξέρετε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο ΟΗΕ σε εθελοντικές ε, συμβολές και ο ΟΗΕ απλώς χρηματοδοτεί το 2% άμεσα το 2%. Το προπολογισμό του ΟΗΕ καλύπτει μονάχα τις ανάγκες του εκπατισμένου προσωπικού που είναι μόνο το 2% του προπολογισμού της ΟΥΡΑ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Θα σταματήσω εδώ και είμαι έτοιμος να απαντήσω τα ερωτήματά σας εάν υπάρχουν και η Φαμπιάν ίσως μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Λιβάνου για να σας δείξω πώς η κρίση της Συρίας επηρέασε και την υπηρεσία. Στο Λίβανο, λοιπόν, έχουμε 270.000 Παλαιστινίους πρόσφυγες. Και ήδη βρίσκονται σε μια πάρα πολύ βάλλοντη κατάσταση. Περιορισμένα δικαιώματα, περιορισμένη πρόσβαση σε δημόσιε υπηρεσίες και ευκαιρίες και ο προϋπολογισμός στο Λίβανο. Ήταν ε, τόσο περιορισμένος που όταν ε, κατέφθασαν ε, οι πρόσφυγες από τη Συρία ήταν κάτι παραπάνω από 40.000. Άρα, τα θέματα για παράδειγμα υγείας και εκπαίδευσης και σχετική νομοθεσία ήταν υπό μεταρρύθμιση. Και προφανώς ε, η άφηξη των ε, μεταναστών είχε αρνητικό αντίκτυπο στις μεταρρυθμίσεις αυτές, γιατί προφανώς ε, έπρεπε να προληφθεί και ένας προπολογισμό για τους μετανάστες από τη Συρία. Υποστηρίζουμε τον UNRWA πέρα από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό σε ό,τι αφορά το Λίβανο και την Ιορδανία, αλλά ιδιαίτερως στο Λίβανο. Και τους υποστηρίζουμε και σε διμερές επίπεδο και μέσω του Ταμείου για την Συρία. Πέρα λοιπόν από το γενικό προϋπολογισμό υποστηρίζουμε την υπηρεσία και μέσω της διμερούς ε, υπηρεσίας και μέσω του ειδικού ταμείου σε ό,τι αφορά το διμερές επίπεδο για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ενίο πλαίσιο υποστηρίξης 2014-2016 χωρίσαμε 10 εκατομμύρια για την UNRWA 5 εκατομμύρια για την, τα καταλήμματα και 5 εκατομμύρια για τα θέματα εκπαίδευση. Χρηματοδοτούμε δε και την υπηρεσία με επιπρόσθετους πόρους για την υποστήριξη προς τον Λίβανο σε ό,τι αφορά την κρίση στη Συρία και έχουμε υποστήριξη 4 εκατομμυρίων για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στα καταλήμματα, στους καταβλισμούς και έχουμε και ένα πρόγραμμα, πρόγραμμα 15 εκατομμύρια το οποίο είναι σε φάση προετοιμασίας, 12 εκατομμύρια για το Λίβανο και 3, 3 εκατομμύρια για την Ιορδανία περίπου προβλέπονται. Επιπροσθέτως, υποστηρίξαμε και την ανοικοδόμηση του καταβλισμού Ναχιλ έξω από την Τρίπολη ένα πρώτο πρόγραμμα 12 εκατομμυρίων χρηματοδοτήθηκε από το εργαλείο της σταθερότητας και της ειρήνης και έχουμε 14,5 εκατομμύρια επίσης τα οποία είναι σε φάση έγκρισης ε, ως χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν και ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, να σας ευχαριστήσω και για όλα τα έγγραφα που μας διαβιβάσατε. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό για μας. Και έχω δύο ερωτήσεις να κάνω. Δεν ξέρω αν και οι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Πείτε μας αν θέλετε ε, εν γέννη ποια είναι η διαφορά της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο Λίβανο και στην Ιορδανία. Είπατε ότι υπάρχουν διαφορές συγκεκριμένες. Πείτε μας κάτι παραπάνω για να ξέρουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς και κάτι άλλο ως ε, πληροφορία που ήθελα να σας ε, ρωτήσω. Από 1η Ιανουαρίου του 2016 άκουσα ότι υπάρχει ε, μία αλλαγή σε ό,τι αφορά το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης που πληρώνεται, που επιστρέφεται από τον άνδρα. Έως τώρα ήταν 100% η χρηματοδότηση αυτή. Τώρα υπάρχει μία συγχρηματοδότηση 5% αν πρόκειται για παλαιστινιακά κρατικά νοσοκομεία και 15%, συγγνώμη, για νοσοκομεία του και 15% είναι, πρόκειται για εθνικά, για κρατικά ε, νοσοκομεία. Ισχύει αυτό. Υπάρχει προπτική να αλλάξει αυτό. Προκαλούνται προβλήματα. Άκουσα ότι γίνονται διαδηλώσει και υπάρχουν ενστάσει. Δώστε μα κάποιε πληροφορίε γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο αυτό. Λοιπόν, η βασική διαφορά μεταξύ Ιορδανία και Λιβάνου είναι η εξή. Στην Ιορδανία περισσότεροι πρόσφυγες έχουν υπηκότητα και έχουν δικαίωμα εργασία, έχουν άδεια εργασία, το οποίο δεν συμβαίνει στον Λίβανο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Γι' αυτό και περισσότεροι πρόσφυγες έχουν καταφύγει στην Ιορδανία, αν και έχουμε μικρότερο προπολογισμό. Όσον αφορά την μεταρρύθμιση στην υγεία, όπως προείπα, η ούνρα ήταν να τροποποιήσει τους κανόνες παροχής υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Όμως, λόγω του αυξημένου πλήθους προσφύγων, και επίσης λόγω των πολιτικών προβλημάτων, λόγω των αντιπαραθέσεων στους καταβλισμούς, ίσως επίσης λόγω και κακής επικοινωνικής πολιτικής και τακτικής όλη Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους δεν ήταν πολύ καλοδεχούμενη αυτή η αλλαγή στα της υγείας. Είχαμε διαδηλώσεις. Δεν έχω ενημερωθεί για τις ε, απολύτως τελευταίες εξελίξεις. Όμως από ό,τι ξέρω, οι αλλαγές έχουν παγώσει και αυτή τη στιγμή τρέχουν συζητήσεις τους καταβλισμούς. Από ό,τι κατάλαβα, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερο. Το σύστημα βεβαίως θα αλλάξει. Όμως δεν εξηγήθηκαν με σαφήνεια οι αλλαγές. Ξέρετε ότι τελευταία είχαμε ταραχές τους καταβλισμούς. Είχαμε μια λίγο εκρηκτική κατάσταση. Είναι και αυτό μία από τις παραπλευρές επιπτώσεις της κρίσης στη Συρία. Ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους καταβλισμούς όπου κρύβονταν τζιχαριστές. Εξαιτία αυτού είχαμε και πολιτικές αντιπαραθέσεις, πολιτικού χαρακτήρα αντιπαραθέσεις στους καταβλισμούς σχετικά με το κατά πόσον τους αφήνουμε ή όχι να μπουν, τους αφήνουμε να βγουν, τι θα κάνει ο στρατός κλπ. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, κάποιοι τέτοιοι τζιχαριστές παραδόθηκαν στα, στις ενοπλές δυνάμεις του Λιβάνου, όμως η κατάσταση είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή. Θα τα ακούσετε βεβαίω με περισσότερε λεπτομέρειε στην Πυρητό. Όχι μόνο λόγω του αυξανωμένου πλήθους των προσφύγων, αλλά και λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Συρία, λόγω της σύραξης εκεί. Υπάρχουν εντάσεις και εντός και στον περίγυρο των καταβλισμών που καθιστούν πολύ, δύσκολες, πολύ δύσκολη την εφαρμογή των αλλαγών που θέλει να εφαρμόσει η UNRWA. Πρόεδρος. Μπουρχαρτ την UNRWA είναι εδώ. Καλώς ήλθατε. Εμείς προετοιμάζουμε την ε, επίσκεψή μας όπως γνωρίζετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πρόσθεσετε κάτι. Δεν ξέρω αν ακούσατε προηγουμένως την ερώτηση, αλλά ακούσατε σίγουρα τι απαντήσει τη Κομισιόν, οπότε αν έχετε κάτι να απαντήσετε παρακαλώ. Ε, μόνο και μόνο για τους σκοπούς της προετοιμασίας μας εν ώψη αυτής της αποστολής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. <clears throat> Δεν θα προσθέσω πολλά. Απλώ θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας για την αποστολή που έχει διοργανώσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσετε να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια την κατάσταση και να δείτε τα προγράμματά μας τα οποία σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χαιρετίζουμε αυτό και θέλω να σας πω, συγγνώμη, καθυστέρησα και δεν, δεν είδα, δεν άκουσα το σύνολο του ερωτήματος. Η μεταρρύθμιση στα υγειονομικά έχει δημιουργήσει πολλά, πολλή αντίδραση σε κάποιο βαθμό. Ο Ματίας Σμάλερ, ο διευθυντής για τα θέματα αυτά, θα έρθει εδώ για, διαπραγμάτευση για διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είναι, έχει γίνει και διευθυντής για την Συρία και θα χρειαστεί να πάει στη Δαμασκό σε λίγο και θα πρέπει να βρούμε ένα αντικαταστάτη του για το Λίβανο, αλλά πάλι θα είναι ακόμα στο Λίβανο όταν βρεθείτε εσείς. Για τη μεταρρύθμιση για τα υγειονομικά θέματα άκουσα κάποιες ε, πληροφορίες που εστάλει στους πρόσφυγες τους Παλαιστίνιους δεν ήταν σαφή τα πράγματα. Εμείς έχουμε μια διαφορετική άποψη. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε αυτή τη μεταρρυθμίση, η οποία είναι και προς το συμφέρον τους, πιστεύω, προς όφελός τους. Υπήρξε όμως μια παρανόηση αυτή της ε, πρότασης και υπήρξε και πολιτική εκμετάλλευση αυτής της παρανόησης, όπως είπαν και οι συνάδελφοι της Κομισιόν. Αυτό μετετράπησε ένα πολιτικό θέμα που δεν έχει να κάνει τόσο με τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης αλλά περισσότερο με τη στάση ορισμένων πολιτικών ε, φορέων έναντι της ε, Ούνρα και εναντίον του, έναντι του Λιβάνου. Και ένα άλλο θέμα είναι η κατάστασή τους στην Ιορδανία. Η δυνατότητα υπηκότητας, ναι, η Ιορδανία ήταν πολύ γενναιόδορη και έδωσε προσωρινή υπηκότητα στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια διαφοροποίηση η Ιορδανία θεωρεί ότι αυτό είναι μια ανθρωπιστική δράση για να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να μπορούν να έχουν ελευθερία διακίνησης μέσα στην Ιορδανία, αλλά αυτό δεν αποτελεί για αυτούς πλήρη ενσωμάτωση, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανασταλεί. Και κάποιοι από εσά το γνωρίζουν αυτό, ότι η προσωρινή υπηκότητα δεν είναι πραγματική υπηκότητα, ακριβώς γιατί μπορεί να ε, αρθεί, να ανασταλεί. Και έχουμε δει και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ότι η Ορδανία έχει μειώσει τον χρόνο ανανέωσης αυτών των διαβατηρίων προσωρινής δηλαδή υπηκότητας από τρία χρόνια κατεβαίνουν στα δύο χρόνια και τώρα <clears throat> δεν δίνουν καν νέα διαβατήρια στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως δυνατότητα πλήρους ενσωμάτωσης των προσφύγων στην Ιορδανία. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και την Κομισιόν και την ΟΝΟΡΑ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο περαιτέρω ερώτημα για την προετοιμασία της ε, αποστολής αυτής. Η επόμενη συνεδρίασή μας ήταν στις 26 Σεπτεμβρίου μετά από το ταξίδι μας στην Ιορδανία και στο Λίβανο και θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας εδώ στην Επιτροπή. Αν υπάρχει κάτι λοιπόν που χρειάζεστε θα επανέλθουμε. Παρά την σημαντική συζήτηση για την ανανέωση των μερών του ελεκτικού συνεδρίου και την ψηφοφορία, νομίζω ότι τελειώσαμε πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε. Κάτι τελευταίο. Η τελευταία μας συνεδρία είναι 26 Σεπτεμβρίου, αλλά η συνεδρίασή μας στις 29 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε. Να το ξέρετε αυτό, ότι δεν θα συνεδριάσουμε στις 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, καλό απόγευμα και καλό βράδυ.